we ready, colleagues? Συνάδελφοι, είστε έτοιμοι. Να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας σύνοδο, παρακαλώ. Το βασικό θέμα για σήμερα είναι οι ψηφοφορίες. Μετά τις πρωινές συζητήσεις, ε, σήμερα το απόγευμα ψηφίζουμε. Δεν κατάφερα να ψηφίσουμε σήμερα το πρωί, λόγω των προσκεκλημένων μας. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Τα σημεία που προβλέπετε σήμερα το απόγευμα. Ελπίζω να έχετε όλες τις κάρτες σας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τι κοινέ διατάξεις για τα ευρωπαϊκά ταμεία όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα. Όπως ανήγγυλα στις 3 Σεπτεμβρίου στην έκτακτη συνοδό η Κομισιόν έχει υιοθετήσει μια νομοθετική πρόταση για να τροποποιήσει τις κοινέ διατάξεις και το σχετικό κανονισμό για αυτές, ούτω ώστε να υπάρξουν εξαιρετικά μέτρα, κατεξαίρεση μέτρα για να βοηθηθεί η Ελλάδα. Η Κομισιόν ε, στην έκτατη συνεδρίασή μας παρουσίασε την πρότασή της και λήφθη απόφαση επί της αρχής που υποστηρίχθηκε από όλες τις ομάδες να προσαρμόσουμε την πρόταση και να περάσουμε στο άρθρο 51 απλουστευμένη διαδικασία του ιστορικού κανονισμού μπορούμε να πάρουμε απόφαση επί της αρχής. Ε, δεν μπορούσαμε στις 3 Σεπτεμβρίου γιατί ο Πρόεδρος δεν μπορούσε επίσημα να περάσει από την Επιτροπή μας την Ολομέλεια το θέμα αυτό. Αλλά τώρα έχει πάει το θέμα στην Ολομέλεια και οι τρεις επιτροπές, ε, το ε, απασχόληση και αλία, ε, που έπρεπε να χρηματοδοτήσουν, το έχουν κάνει. Επομένως θα περάσουμε στην απλουστευμένη διαδικασία. Τέλος, χθε έλαβα μια επιστολή από τον πρόεδρο του Κορεπέρ που επιβεβαιώνει ότι το Συμβούλιο αποφάσισε επίση να εγκρίνει την πρόταση τη Κομισιόν χωρί τροπολογίες. Θα ήθελα εσεί σήμερα να, να επιβεβαιώσετε και επίσημα και τυπικά να εφαρμόσουμε το άρθρο 51, ούτω ώστε να παρουσιάσουμε στην πρώτη Ολομέλεια του Οκτωβρίου εκ μέρου τη επιτροπή μα, μία έκθεση που θα εγκρίνει την πρόταση τη Επιτροπή και θα την αλλάζει. Ο κύριος ε, Το υποστηρίζει. Το υποστηρίζετε όλοι. Ευχαριστώ. Έχουμε και την ε, επίσημη απόφαση. Αρκεί αυτό για τη γραμματεία. Ήταν θέμα τυπικό. Και πρέπει να ρωτήσω, υπάρχουν αντιρρήσει. Όχι, δεν υπάρχουν. Ο κ. Μπρουερ απέχει. Όπως και την προηγούμενη φορά. Σας ευχαριστώ όλους. Συνεχίζουμε. Με το επόμενο σημείο, την έκθεση του κύριου Πλάνκο Λόπεθ, τα Ευρωπαϊκά Διαστατικά Ταμεία και Ταμεία Επενδύσεων και η Χρηστή Οικονομική Διακυβέρνηση, κατευθυντήρες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Έχετε τον κατάλογο ψηφοφορίες. Ξεκινάμε με το συμβιβασμό, με τους συμβιβασμού. Συμβασμό 20, παράγραφος 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Πάμε στην ε, πρόταση 1 για τον προπολογισμό. Suggestion 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 4. Για την παράγραφο 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Περνάμε τώρα στο συμβασμό 5 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 38, πρώτο τμήμα. Υιοθετήσαμε το συμβασμό 5, έτσι, μόλις τώρα. Επομένως, καταπίπτει. Καταπίπτουν οι επόμενες, γιατί πάμε στην 38, τροπολογία 38, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβασμός 6, υπέρ, κατά, άποχες, Υιοθετείτε. Συνδεσμός 8. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Συνδεσμός 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 53. Με προφορική τροπολογία. Υπάρχει κάποιος κατά της προφορικής τροπολογίας. Όχι. Ψηφίζουμε την 53 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 54. Τροπολογία 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 56. Περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβιβασμός 59. Ε, τροπολογία 59, πρώτο τμήμα. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 60, τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 9. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Υθετείτε. Συμβασμό 18. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 10. Σε τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά, άποχες, υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Τροπολογία ή μάλλον πρόταση 4 από την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Πρόταση 4. Υπόδειξη 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Συμβιβασμός 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Τροπολογία 81. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός. Όχι, τροπολογία 82. Τροπολογία 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά το ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 82. Ψηφίζουμε τώρα. Δουλεύει. Ψηφίζουμε τώρα. Μια ανοιχτή ψηφοφορία ακόμα. Πέρας πληροφορίας. Απορρίπτεται. Με 29 ψήφους κατά. Σαφέστατο. Συμβασμός 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Συμβασμός 14. Σωστό. Ναι υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. συμβασμός 16 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. συμβασμός 22 να τον βρω πρώτα υπέρ κατά εποχές υιοθετείται συμβασμός 17 υπέρ κατά εποχές υιοθετείται συμβιβασμός 19 υπέρ κατά εποχές υιοθετείται τροπολογία 106 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται τροπολογία 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται υπόδειξη 7 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά εποχές Υιοθετείτε. Τροπολογία 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 117. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Τροπολογία 123. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πρόταση υπό, παύλα υπόδειξη της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η υπόδειξη 9. Θα τη τσεκάρουμε. Α, τσεκάρουμε την 123. Όχι, συγγνώμη, διορθώνει πρόεδρος. Της, την πρόταση 9 της Επιτροπής Προπολογισμών ελέγχουμε τώρα ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 17 ψήφους υπέρ και 21 κατά. Συν μία ακόμα από τους σοσιαλιστές. Παρακαλώ ελέγξτε τον αριθμό των ευρωβουλευτών που ψηφίζουν. Ομάδα σας. Απορρίπτεται πάντως η πρόταση 9. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συνδεσμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές Υιοθετείτε. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 13, παρακαλώ. Ψηφίστε τώρα. Πέρα ψηφοφορίας. Έχουμε ένα παραπάνω βουλευτή από το ΕΛΚ που ψηφίζει αυτή τη στιγμή. να ελέγχεται. Επαναλαμβάνουμε. Ψηφίστε τώρα τη 13. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. Ευχαριστώ. Συμβασμός 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογή 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα ψηφίζουμε ολόκληρη την έκθεση ηλεκτρονικά ψηφίστε τώρα δεν είναι ανοιχτό το σύστημα δεν έχει ανοίξει ψηφοφορία. Ή έχει ανοίξει, ψηφίστε τώρα παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Η έκθεση υιοθετείται. ...28 υπέρ και τα υπόλοιπα νούμερα τα βλέπετε. Να μην τα λέω. Συγχαρητήρια, κύριε Μπλάνκο Λόπεθ. Thank you, Thank you very much. Uh, η επόμενη έκθεση είναι η έκθεση Φερνάντο Ρούας Πολιτική συνοχή και αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Αρχίζουμε με τη συμβαστική τροπολογία 7 στην παράγραφο 1. Υπέρ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 Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 90 με την προφορική. Είναι κανείς κατά της προφορικής, όχι, καλός. Συνεπώς, ψηφίζουμε την τροπολογία με την προφορική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 92. 93 διορθώνει η πρόεδρος. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγξουμε καλύτερα. Α, όχι, όχι, δεν έπρεπε να την ψηφίσουμε την 97 γιατί εγκρίναμε την 29. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ακυρώνεται αυτή η ψηφοφορία δηλαδή, δικό μου λάθος. Πάμε στη συμβαστική 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 108 τροπολογία τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 18. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 19. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 20. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 21. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 23. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 148. όχι 158 που είναι γλωσσική. Άρα πάμε στη συμβαστική 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 171 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 172 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 188. Έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 190 τότε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμός 1 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική αριθμός 1. Συνεδρική σκέψη α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Είναι γλωσσική. Τροπολογία 12 τότε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Στην σκέψη Β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17 είναι γλωσσική, άρα πάμε στη συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Πέρα τη ψηφοφορία. Όχι, δεν έληξε η ψηφοφορία γιατί μένουν ακόμα κάποιοι να ψηφίσουν. Περιμένουμε. Τώρα πέρα τη ψηφοφορία. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, κύριε Здравейте. The next, Επόμενη ψηφοφορία είναι για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2015. Ε, συγητής Ίσκρα Μιχαλιώβα. Συγγήτρια και έχουμε και τον κατάλογο ψηφοφοριών. Ψήφι υπέρ για το τροπολογία 1. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία υπαριθμών 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Η ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία συμβαστική μάλλον 3 υπέρ. Κατά. Αποχές αυτή εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και αυτή υπαριθμών 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 21 εκπίπτει αυτή γιατί εγκρίθηκε η παριθμονή 20 Α, 21 την ψηφίζει πρόεδρος υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Α, αυτή εκπίπτει λοιπόν, ναι, ναι, για αυτά που λέγαμε. Η συμβαστική υπαριθμών 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή τώρα στο σύνολό της η ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει η ψηφοφορία παρακαλώ ψηφίστε ψηφίσατε πέρας και η γνωμοδότηση ενεκρίθη και σας ευχαριστώ πολύ. Ας συνεχίσουμε. με το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το έτος 2016 όλα τα τμήματα. Πρόκειται για γνωμοδότηση που έχει συντάξει η κυρία Σπυράκη. Αρχίζουμε με το συμβαστικό κείμενο, συμβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές ας κάνουμε επαλήθευση σας παρακαλώ ηλεκτρονικά λοιπόν την τροπολογία υπαριθμών 11 αρχίζει η ψηφοφορία παρακαλώ ψηφίστε ψηφίσατε πέρας Εγκρίνεται λοιπόν, αν ε, τα βλέπω καλά. Τροπολογία 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 16. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται αυτή. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εδώ χρειάζεται επαλήθευση ηλεκτρονικά αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ ψηφίστε πέρας η παριθμόν 22. Η παριθμόν 23 τώρα τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές εδώ χρειάζεται παρήθευση Η ηλεκτρονική παρήθευση λοιπόν τροπολογία 24 ψηφίζεται ηλεκτρονικά. Πέρας. Και βλέπετε και στον πίνακα ότι εγκρίθηκε. Τώρα, η ηλεκτρονική ψηφοφορία στο σύνολο της νομοδοτήσεως. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίστε τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση στο σύνολό τη και συγχαρητήρια στην κυρία Σπυράκη. Και τώρα προχωρώ στην ψηφοφορία για την ε, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή της Αδριατικής. Αρχικός συζητητής ο κύριος Ιακοφτσίτση. Χρειαζόμαστε σχόλια. Κύριε Σας ευχαριστώ για όλους όσους συνεργαστήκατε μαζί μου σε αυτή την έκθεση. Πριν από 10 χρόνια δημιουργήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση Αδριατικής ε, Ιωνίου. Εγώ είμαι πρόεδρος. 10 χρόνια μετά έχουμε την πρώτη έκθεση εδώ στο Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι θα πάει καλά η ψηφοφορία και το αποτέλεσμα θα είναι ευνοϊκό. Ευχαριστώ. Περνάμε στην ψηφοφορία. Συμβιβασμό 4. Συμβαστική πρόταση 4. Υπέρ, κατά, αποχέ. Υιοθετείτε. Τροπολογία 27. Υπέρ, κατά, αποχέ. Υιοθετείτε. Συμβασμό 5 υπέρ, κατά, αποχέ, υιοθετείται. Συμβασμό 6 υπέρ, κατά, αποχέ, υιοθετείται. Συμβασμό 8 υπέρ, κατά, αποχέ, υιοθετείται. Τροπολογία 37. We have an oral amendment. Έχουμε και προφορική τροπολογία. Όποιος δεν οποιοδήποτε είναι κατά της προφορικής τροπολογίας θα μιλήσει τώρα. Δεν υπάρχει. Άρα ψηφίζουμε 37 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εποχές. υιοθετείτε. Συμβασμός 7. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Άφετ 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Την 47. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά. Πέρας προφορίας. Απορρίπτεται. Συμβασμός 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Συμβασμός 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Τροπολογία 55. Μία προφορική επίσης τροπολογία. Κάποιος κατά. Όχι. Ψηφίζουμε την 55 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 57 υπέρ Καταπίπτει. Συγγνώμη. συμβασμό 12. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Υιοθετείτε. 58. Τροπολογία 58. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Υιοθετείτε. Συμβασμό 13. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται συμβασμός 14 Περ. κατά εποχές υιοθετείται τροπολογία 70 Περ. κατά εποχές υιοθετείται συμβασμό 41 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται ΑΦΕΤ 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Την ΑΦΕΤ 10. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. 77, τροπολογία 77, υπέρ. Κατά. Εποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 77. Ψηφίζουμε. Πέρας φοφορίας. Υιοθετείτε. Τροπολογία 79. Υπέρ κατά αποχές πρέπει να τη ελέγχουμε την τροπολογία 99 με ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίστε τώρα πέρας της ψηφοφορίας υιοθετείτε συμβασμός 15 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε Συνδεσμός 38 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε χρονικά. Την τροπολογία 87 έναρξη της ψηφοφορίας πέρας υιοθετείται. 87. Συμβασμός 16 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Τροπολογία 98 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Τροπολογία 99 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι υιοθετείτε. Τροπολογία 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείτε. 108. Υπέρ. Έχουμε και ένα συμβασμό. Το συμβασμό 17. Συγγνώμη. Συμβασμό 17 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Υιοθετείται. Τροπολογία 108 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Υιοθετείται. Τροπολογία 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 111. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. MV2 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται νομίζω Θέλω να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τώρα την MV2 ηλεκτρονικά Πέρα τι ψηφοφορίας υιοθετείται Πες 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ. Σηκώστε τα χέρια σας όμως. Γιατί πες 22 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 117 υπέρ κατά άποχες υιοθετείτε. 118 υπέρ κατά άποχες υιοθετείτε. 120 υπέρ κατά άποχες υιοθετείτε. 121 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 122 υπέρ κατά εποχές διαθετείτε 123 υπέρ κατά αποχές Κατόν 124 υπέρ κατά εποχές διαθετείται Συμβασμός 18 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Εύη 12 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι υιοθετείται. Πες 14 υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την ΠΕΣ 14. Ψηφίζεται τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Τροπολογία 133. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Πες ή. Πες 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πες 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Πες 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Συμβασμό Συμβασμός 19. Περ. Κατά. εποχέ. Υιοθετείτε. 137 υπέρ. Κατά. εποχές Υιοθετείτε. Συμβασμός 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Πες 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε χρονικά την πες 12. Ψηφίτε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Εκατόν σαράντα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Yeah. You want to check. Okay. Θα το τσεκάρουμε. Ναι. Ξαναψηφίσουμε στον την 142. Πέρας φοφορίας.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 Υιοθετείται η τροπολογία 143. Πες 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. MV10 υπέρ κατά εποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά την MV10 ψηφίστε τώρα πέρας φοφορίας απορρίπτεται πέσω 17 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. MV19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πες 23 υπέρ καταπίπτει. Ψηφίζουμε την ΠΕΣ 23 υπέρ κατά Αποχές ελέγχουμε χρονικά. Ψηφίστε τώρα. Πέρας φοφορίας. Υιοθετείτε. Συμβασμός 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. Συμβασμός 22. Κατά. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε MV 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται MV 27 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά την MV 27 ψηφίστε τώρα Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Συμβασμός 23. Υπέρ. Κατά. Κα... Αποχές υιοθετείτε. Συμβασμός 24. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα του συμβασμού 24 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα του Συμβασμού 24 ηλεκτρονικά. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα του Συμβασμού 24. υπέρ κατά αποχές Συνδεσμός 25 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Υφετείτε. δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβασμός 40 υπέρ κατά άποχες υιοθετείται. Συμβασμός 26 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 183 υπέρ κατά αποχές Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 183. Ψηφίζω τώρα. The vote is closed. Υιοθετείτε. Συμβιβασμός 27. Σε δύο τμήματα. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Παρακαλώ ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 192 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 200 200 εδώ είναι η ψήφη υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απερίφθη τροπολογία 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πες 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 205 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ένβη υπάρχει μόνο 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 210 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πες 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία παθών 216 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ένβι 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πες 19 υπέρ κατά αποχές εδώ χρειάζεται επαλήθευση πες 19 η ηλεκτρονική ψηφοφορία για επαλήθευση αρχίζει ψηφίστε παρακαλώ πέρας και απορρίπτεται. Συμβιβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πες 13 υπέρ κατά αποχές αυτή νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά χρειάζεται επαλήθευση καταλαβαίνω ναι πες 13 λοιπόν ηλεκτρονική ψηφοφορία Πέρας. Μάλιστα εγκρίθηκε λοιπόν. Η 13 πες. Τροπολογία 219 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 220 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. 221 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 222 υπέρ κατά αποχές αυτή εγκρίνεται συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 224 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 225 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 226 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτή συμβιβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 232 σωστό 232 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 235 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πηγαίνουμε τώρα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος 21, NV21, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 240 με χωριστή, με, δηλαδή ψηφορία κατά τμήματα, σε δύο τμήματα, την οποία έχει ζητήσει ο κύριος Γιάκοφτσιτς της και την έχει διανύμει κιόλα σε όλα τα μέλη. Την δέχεστε, δέχεστε να γίνει η ψηφοφορία κατά τμήματα. Ωραία. Πρώτο τμήμα της ψηφού, ψήφι πέρα. Κατά, αποχές. Ας κάνουμε επαληθευσή Πρόκειται για την τροπολογία 240, πρώτο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. Το δεύτερο τμήμα του 240 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εδώ νομίζω ότι απορρίπτεται. απορρίπτεται λέτε. Μάλιστα απορρίπτεται. 241 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 242 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπαριθμών 247 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 248 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 249 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτή 250. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 251. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή. 252. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 253. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 254 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 263 ψήφι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται 265 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτό 266 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 267 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 268 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έρχομαι τώρα στα εκτιμώντα, δηλαδή τι αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αυτή. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένβη 2 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται αυτή. NV3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές. Εδώ χρειάζεται επαλήθευση. Τροπολογία 12 λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας. Και όντως εγκρίθηκε. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αυτή τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σι, υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε, θα παληθεύσουμε για την ε, πες αλίας Συ. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πες D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πες F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πες H. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πες I. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πες J υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πες K υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πες L υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πες M υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της φοφορίας. Εγκρίθηκε η έκθεση. Συγχαρητήρια κύριε Γιάκοβιτς. Έχω κάποια θέματα ακόμα που θα ήθελα να συζητήσουμε. Πριν τελειώσουμε τη συνεδρίαση δηλαδή, πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι έχετε πάρει την περίληψη των αποφάσεων των συντονιστών που συνεδρίασαν σήμερα το πρωί. Συμφωνείτε? εγκρίνετε. Ωραία. Διάφορα. Υπάρχει τίποτα στα διάφορα παρακαλώ. Όχι. Καλώς. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα λάβει χώρα στις 15 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ όλους. Έληξε συνεδρίαση.